Σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 6 του κανονισμού, ο πρόεδρος της διάσκεψης των πρόεδρων των επιτροπών με ενημέρωσε ότι δεν υπήρξε καμία αντίρρηση από την διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών στη σύσταση της Επιτροπής Αλίας να μην εναντιωθεί σε μια κατεξοδότηση πράξη. Αν μέσα σε 24 ώρες καμία πολιτική ομάδα ή αν δεν υπάρξει ελάχιστος αριθμός ευρωβουλευτών που να προβεί σε αντιρρήσει, τότε η σύσταση αυτή θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται. Στην αντίθετη περίπτωση, η σύσταση αυτή θα υποβληθεί στη διαδικασία ψηφοφορία. Η σύσταση αυτή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας.